Σήμερα το πρωί αρχίζουμε με το σημείο 13 της ημερήσιας διάταξης μια νέα ψηφιακή στρατηγική για την Ευρώπη. Θα πρότεινα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν για να μας δώσει, να μας κάνει μια κάποια εισαγωγή. Τον παρακαλώ συγχρόνως να είναι σύντομο για να μπορέσουμε μέχρι το μεσημέρι να έχουμε τελειώσει τα θέματα της σημερινής διάταξης. Παρακαλώ κύριε του έχετε το λόγο. Okay, thank you, Mr. President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σήμερα το πρωί να σας πω ότι μπορώ από πλευράς ενημέρωσης για το πώς έχουμε προχωρήσει μέχρι σήμερα όσον αφορά το θέμα μας. Ο κύριος Μπαρόσο, όπως ξέρετε, έχει τάξει αυτό το θέμα ως ύψη προτεραιότητα για το όραμα του για το 2020 και είχε προβεί στις 3 Σεπτεμβρίου και σχετική αναγέννηση προς το Κοινοβούλιο τότε που είχε ανακοινώσει κατευθύνες γραμμές της πολιτικής του και είχε πει επιλέξει ότι η επομένη επιτροπή πρόκειται να εκπονήσει μια τέτοια ψηφιακή ατζέντα και ότι θα υπάρξει ένα αντίστοιχο νομοθετικό πρόγραμμα ώστε να αρθούν οι σχετικοί φραγμοί για να έχουμε μια τέτοια αυθεντική ενιαία ψηφιακή αγορά και θα προωθήσει τις επενδύσεις ε, μέσω του διαδικτύου και να σταματήσει να υπάρχει χάσμα και κενό γιατί όλο ένα και περισσότερο σημαντικό είναι αυτό, η συμμετοχή του Ιντερνετ στην ανάπτυξη τη οικονομία. θα πρέπει να έχουμε ασφάλεια στα δίκτυα και αυτό επίση θα το φροντίσουμε. Επομένως, περίπου αυτά είπε σε εκείνες οι καθητήρες γραμμές και στι 24 συνδικά την περασμένη εβδομάδα ε, ενέκρινε η Επιτροπή αυτό το έγγραφο για διαβούλευση, το οποίο αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2020, όπου μπορείτε να δείτε ε, αυτήν την ψηφιακή ε, ατζέντα που ε, μνημονεύεται σε διαφορετικά σημεία αυτού του κειμένου και βλέπετε για αυτή την ενιαία αγορά για το διαδίκτυο μπορεί να δείτε επίσης το πόσο θεωρούμε θα πρέπει η οικονομία να στηριχτεί στο διαδίκτυο να προχωρήσουμε προς ε, καινοτομία, προς ε, καινούργια μορφή υπαρχής υπηρεσιών, συμμετοχή, ελευθερία έκφρασης για τον κόσμο. Οπότε, μέχρι τις 15 πρώτου θα συνεχιστεί η διαβούλευση με βάση αυτό το έγγραφο και η Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνέχεια θα εκπονήσει ένα έγγραφο το οποίο θα υποβληθεί στο Ειρηνό Συμβούλιο και ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά και θα εγκριθεί τον ε, Μάρτιο του χρόνου. η Γενική Διεύθυνση για την κοινωνία της πληροφορίας και τα μέσα έχει προχωρήσει στη δουλειά της και χαιρετίζουμε επομένω την παγίωση αυτής της ψηφικής ατζέντα που θα είναι αρμοδιότητα της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης και στην καινούργια Ευρωπαϊκή Επιτροπή οπότε και θα έχουμε κάποιες ε, μελέτες θα προχωρήσει η διαβούλευση και να χαράξουμε τη νέα στρατηγική που θα αφορά την ψηφιακή ατζέντα. Τώρα, να σας πω τα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης που ξεκίνησε στις 4 Αυγούστου ε, μέχρι τις 9 ε, Οκτωβρίου. 834 απαντήσεις πήραμε ε, μέσω του διαδικτύου και 150 ε, εγγράφους όσον αφορά το ερωτηματολογείο μας. Επεξεργαζόμαστε αυτά τα ερωτηματολόγια και πρόκειται να δημοσιεύσουμε σύντομα μία σύνοψη. Θέλουμε τώρα να δούμε από ποσοτικής πλευράς τα αποτελέσματα και Εσείς θα ενημερωθείτε επίσης 92% των όσων απάντησαν είπαν ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η στρατηγική αυτή της ε, ψηφιακής διάστασης και ως ύψιστη προτεραιότητα είπαν όσοι απάντησαν ότι είναι το πώς θα έχουμε υψηλές ταχύτητες στο διαδίκτυο και ανοιχτά δίκτυα. Δεύτερη τώρα προτεραιότητα για όλους, το οποίο κάπως μας εξέπληξε περισσότερο, είναι το θα πρέπει να υπάρχει έρευνα, καινοτομία και άλλες προτεραιότητες είναι η ενιαία online αγορά. Από επτά διαφορετικά θέματα και εκτό από αυτά τα τρία κορυφαία, στη τέταρτη θέση ήταν τα θέματα τα οποία αφορούν το πώς θα γίνει η μετάβαση σε μια οικονομία ενεργειακής αποτελεσματικότητας με, χαμηλή, ε, με χαμηλέ εκπομπές άνθρακα ή διοξιδίου του άνθρακα. Τώρα, 65% ήταν, από φυσικά πρόσωπα και άλλες από φόρες και τα φυσικά πρόσωπα προτίμησαν να τονίσουν το θέμα των δικαιωμάτων των χρηστών, ποιότητα ζωής, ενώ οι φορείς, τα νομικά πρόσωπα, οι εταιρείε ε, τόνισαν ζητήματα τα οποία αφορούν έρευνα και καινοτομία. Απασχόλησε. Και επίσης ε, θα πρέπει να υπάρξει νέα στρατηγική για ανοιχτά δίκτυα και τα νομικά πρόσωπα κυρίως θέλουν να υπάρχουν κάποια προγράμματα με μετρήσιμους στόχους που να επιδέχονται αξιολόγηση μακροπρόθεσμα. Αυτή είναι η ανοιχτή διάσταση πάντοτε προέκυπτε από το 90% των απαντήσεων ανοιχτό ίντερνετ, ανοιχτά πρότυπα επομένως το να είναι ανοιχτά αυτός ο χαρακτηρισμός ε, κυριάρχησε και 90% δεν σημαίνει βέβαια ότι ήταν μόνο τα φυσικά πρόσωπα αλλά και τα νομικά πρόσωπα αυτό ετώνησαν. Έργα υποδομής για το μέλλον και αυτό έχει σημασία και εμείς ρωτήσαμε κατά πόσο θα πρέπει να έχουμε δημόσιες επενδύσεις όσον αφορά ε, τα έργα υποδομής που απαιτούν έργο πολιτικού μηχανικού και 78% μας είπαν ότι είναι υπέρ του να αναζητηθούν τρόποι ούτως ώστε να έχουμε συνέργεια στις επενδύσεις για τις υποδομές και να είναι κυρίαρχος ο δημόσιος τομέας σε αυτό. Ρωτήσαμε και για το ψηφιακό περιεχόμενο όσον αφορά αυτό το ερωτηματολόγιο που τους υποβάλαμε online και εν προκειμένου διαπιστώθηκε ότι 79% ήταν υπέρ του να υπάρχει το δικαίωμα στο περιεχόμενο σε πολλαπλές πλατφόρμες και το οποίο να κατοχυρωθεί υποτύπων δικαιώματο που προκύπτει από κάποιο είδου καταστατικό χάρτη δικαιωμάτων για τα φυσικά πρόσωπα, επίσης δικαίωμα στην ιδιωτικό βίο, ουδετερότητα, παγκοσμιότητα στην κάλυψη, ουδετερότητα και 75% από όσων απάντησαν είπαν ότι θέλουν να υπάρχει κάποιο είδου ε, ε, νομική βάση γι' αυτά και 61% είπαν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια εναρμονισμένη ενωσιακή ε, προσέγγιση 49% θέλανε να υπάρχει κάποιο άλλο είδους ε, ε, νομική βάση, βάση του εθνικού δικαίου ή κάπω αλλιώ. Και θέματα τα σχετικά με έρευνα θα πρέπει να τα αναφέρουμε δύο λίγο. Όταν ρωτήσαμε για έρευνα και καινοτομία πού είναι πιο καλή η Ευρώπη, μας απάντησαν ότι οι τέσσερις κορυφαίοι τομείς είναι η ενέργεια και το περιβάλλον, σχετικές τεχνολογίες, η τεχνολογία σχετικά με την υγεία, παιδεία, πολιτισμός και τα δίκτυα. Με αυτή την σειρά που σας τα αναφέρω. Και όταν ρωτήσαμε ποιοι είναι οι τομείς που έχουν στρατηγική σημασία, μας είπαν ότι είναι η ενέργεια, το περιβάλλον, ε, παιδεία και πολιτισμός, αλλά όσον αφορά το software και υπηρεσίες δικτύου, μας είπαν ότι δεν είμαστε τόσο καλοί αλλά θεωρούνται από του απαντήσαντες ότι είναι πάρα πολύ σημαντική τομή. Τα ξέραμε αυτά. Οι ε, υπηρεσίε δικτύου, η νανοτεχνολογία, μικροτεχνολογία, ε, οι τηλεπικοινωνίε. και γενικά προέκυπτε από αυτό το κομμάτι του δημοτολογίου ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προσπαθήσει περισσότερο όσον αφορά την έρευνα την ε, καινοτομία και να υπάρξουν ε, μέτρα. Και θα πρέπει να δουλέψουμε μέσα από τα διαρροτικά ταμεία και το πρόγραμμα πλαίσιο για την ε, έρευνα. Πάρα πολύ έντονα ενδιαφέρθηκαν οι απαντήσαντες για το πρωτογενές και δευτερογενές δίκαιο το οποίο θα περιχαρακώσει την καινοτομία και την ανάπτυξη στην Ευρώπη ε, επί τη βάση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Και, εν κατακλείδη, όσον αφορά αυτήν την ε, δημόσια διαβούλευση, τα αποτελέσματά της, όσον αφορά τις δημόσιες online υπηρεσίες θα γνωρίζετε ότι στα προηγούμενα δύο στατηγικά προγράμματα πλαίσια ε, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας επίσης προβλήθηκαν και σε 73% από όσους απάντησαν είπαν ότι βασικός μέσο όπου θα πρέπει να προσπαθήσουμε είναι η διαφάνεια αυτών των υπηρεσιών. Και άλλοι τόσοι είπαν ότι θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος όσον αφορά το τι πληροφορίες τροφοδοτούν την παροχή αυτών των πληροφοριών γιατί δεν θα πρέπει να υπάρξει ε, υπερβολική, καταχρηστική, παράνομη χρήση των δεδομένων των πληροφοριών από κυβερνητικούς φορείς, από δημόσιες αρχές κλπ τελευταίο που θέλω να σας αναφέρω όσον αφορά το πώς θα πάμε σε μια ε, οικονομία χαμηλών ε, εκπομπών άνθρακα πρόκυψε ότι πολλοί απάντησαν σε αυτό το κομμάτι του ερωτηματολόγιου και βγήκε πως τα φυσικά πρόσωπα που απάντησαν είπαν ότι προβληματίζονται γιατί δεν υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές ούτως ώστε ο κόσμος να μπορεί να αλλάξει τη συμπεριφορά του αλλά και τα νομικά πρόσωπα προβληματίζονται γιατί ότι δεν ξέρουμε για εναλλακτικά ε, επαγγελματικά επιχειρηματικά μοντέλα για αλλαγή στον τρόπο ζωής άρα είπαν ότι αυτό θα πρέπει να προσέξουμε και όχι τόσο την, ε, τη δράση μέσω της ε, νομοθεσίας και δεσμευτικών ρυθμίσεων. Τι να πούμε πριν να λάβει ο καινούριο επίτροπο. Βεβαίω και το αποτελεσματικό του ερωτηματολογίου πρόκειται να τροφοδοτήσει το έργο μα σε συνέχεια του εγγράφου του 24 Νοεμβρίου για την ε, διαβούλευση εν ώψη ε, της δουλειάς του Ιανουαρίου και μάλλον θα έχουμε κάποιο είδους έγγραφο εργασία το οποίο πρόκειται να δημοσιευθεί μάλλον παράλληλα με το έγγραφο που θα αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020. Και όλη η Επιτροπή από κοινού θα ασχοληθεί με την ψηφιακή Ευρώπη, με αυτή την ατζέντα του, του χρόνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Θα δώσω το λόγο όμω στην εισηγήτρια την κυρία Καστίγιο. Sí, eh, muchas gracias, eh, presidente. Eh, muchas gracias a la Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήρθε σήμερα εδώ και μας ε, εξέθεσε το περιεχόμενο τη στρατηγικής της ψηφιακής για την Ευρώπη. Από ό,τι φαίνεται, λόγω της συγκυρίας στην οποία βρισκόμαστε εν ώψη δηλαδή της συγκρότησης της καινούργιας επιτροπής θα πρέπει να περιμένουμε όμως ο πρώτος Μπαρόσο ξεκάθαρα τόνισε ότι αυτός ο ψηφιακός προσανατολισμός αυτή η ψηφιακή στρατηγική είναι η πιο σημαντική στρατηγική που θα διαπνέει, που θα κανονίσει, που θα ρυθμίσει όλες του τις κινήσεις και θα έρθει εδώ να μας τα πει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα. Εγώ θέλω να σας πω το εξή. Ε, ευτυχώς σήμερα από πολλές κατευθύνσεις πάμε προς τον ίδιο στόχο. Δηλαδή το πώς θα βρούμε αυτήν την ψηφιακή ατζέντα. Έχουμε δηλαδή κάποιου ιδιωτικού φορεί που ήδη έχουν προχωρήσει προ τα εκεί. Επίση, επ' αυτού δούλεψε η Σουηδική Προεδρία. τώρα θα το ξεκινήσει το ίδιο η Ισπανική Προεδρία, φυσικά η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο επίσης ανέλαβε εκθεσίδια πρωτοβουλίας. Οπότε και εγώ ανέλαβα ένα τέτοιο κείμενο, βρίσκομαι στη φάση του σχεδίου κειμένου θα ζητηθεί αρχές του Ιανουαρίου. Και έτσι ελπίζουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι έγκαιρα όταν έρθει η ώρα να καθορίσει η Κομισιόν και να ε, παρουσιάσει και να ανακοίνωσή της για την ε, ε, ψηφιακή ατζέντα. Απρίλιο ή Μάιο. Ελπίζουμε ότι τότε θα μπορέσουμε να έχουμε μια ξεκαθαρή θέση. Και θα μπορέσει η Κομισιόν να χρησιμοποιήσει τη δική μας θέση. Οπότε, να μπορέσουμε έγκαιρα να συμμετάσχουμε σε μια τέτοια προβληματική. Όταν τρία θεσμικά όργανα, οι προεδρίες, οι ιδιωτικοί φορείς, ε, νομικά πρόσωπα. Όλοι, όλοι, όλοι να έχουν συνειδητοποιήσει ότι βαδίζουμε προς τη διαμόρφωση μιας ε, ψηφιακής, ανοιχτής και ανταγωνιστικής αγοράς. Άρα δεν θέλουμε πισωγυρίσματα και από αυτής της πλευράς το Κοινοβούλιο πιστεύω ότι υπάρχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο θα πρέπει να προσέξει, να είναι κάτι σαν αφετηρία, σαν θεμέλιο για αυτή τη στρατηγική. Δηλαδή, ότι έχουμε τώρα μια επανάσταση στις τηλεπικοινωνίες. Δηλαδή, την ψηφιακότητα, την ψηφιακή διάσταση. Αλλά αυτό όμως είναι κάτι το οποίο το, το, το, το παίρνουν στην πλάτη τους, το αναλαμβάνουν τα πρόσωπα, οι άνθρωποι. Είναι κάτι το οποίο αφορά το σύνολο του πληθυσμού, όλους. Και αν δεν γίνει κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν ποτέ να φτάσουμε σε αίσιο πέρας. Διότι αντίθετα από άλλες ε, ιστορικές στιγμές, από άλλα γεγονότα, ε, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να πετύχουμε την ψηφιοποίηση και όλοι να μπορέσουν να συμμετάσχουν και να επέμβουν. Όχι κάποιες ελίτ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και έτσι λοιπόν από τη βάση προς τα πάνω να υπάρξει τέτοιου είδου ολοκληρωμένη αντιμετώπιση από όλους. Βεβαίως και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αποτελέσματα για τα αποτελέσματα τα οποία μας είπατε κύριε εκπρόσωπε της ε, Κομισιόν. Ε, ξέρω ότι ακόμα ψεργάζεστε αυτά τα στοιχεία και τα αναλύετε, αλλά να κάτσουμε να λάβουμε υπόψη το χρονοδιάγραμμα. Ε, έχουμε τμηματικά αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά όμως είναι πάρα πολύ χρήσιμο τόσο μας είπατε. Ευχαριστούμε για την εισήγησή σας και αρχίζει τώρα αυτός ο προβληματισμός που κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σημαντικός για να μπορέσουμε να περιχαραγώσουμε, να καθορίσουμε τις στρατηγικές, τους στόχους ε, γιατί πρόκειται για μια ευκαιρία που θα δώσει όθηση στις οικονομίες της Ευρώπης. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την Κομισιόν για την έκθεση που παρουσίασε. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά για την ανταγωνιστικότητα και ε, βεβαίω ε, τα τελευταία χρόνια είναι προτεραιότητά μας ενημέρωση για την ε, ψηφιακή πολιτική αν θέλετε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο θεωρώ ότι η έκθεση είναι λίγο παρά είναι αισιόδοξη. Ε, δεν υπάρχει προφανής σύγκριση με τα άλλα μέρη του πλανήτη, με τους ανταγωνιστές μας. Λέμε ότι έγιναν πρόοδοι στην Ευρώπη, αλλά δεν λέμε τι έγιναν αλλού. Βεβαίως έγιναν θετικά πράγματα την περασμένη πενταετία. Παρόλα αυτά καθίστε, υστερούμε σε σχέση με άλλες περιφέρειες, περιοχές του κόσμου. Θα ήθελα η ψηφιακή ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ήταν πολύ πιο φιλόδοξη από ό,τι ήταν την τελευταία πενταετία. Πιο συγκεκριμένοι στόχοι πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα για το τι θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει στην Ευρώπη μελλοντικά. Μιλάμε για τον αριθμό των χρηστών του διαδικτύου. Στην έκθεση της Κομισιόν μιλάει για 43% το 2005 που ανέβηκε το ποσοστό αυτό στο 56% στο 2008 είναι θετική εξέλιξη αλλά είναι επαρκές να έχουμε μόνο το μισό πληθυσμό της Ευρώπης που χρησιμοποιεί διαδίκτυο η δυναμική, το ποσοστό μπορεί να είναι μεγαλύτερο από άλλες χώρες αλλά η δυναμική είναι πιο αργή στην Ευρώπη και φοβούμε ότι αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό στο μέλλον θα είμαστε πίσω από κάποιες άλλες χώρες και περιοχές. Τώρα, για την πρόσβαση στις ευρυζωνικές συνθέσεις 2 Mbits ανά δευτερόλεπτο λέμε είναι χαμηλό το κατόφλι αυτό αν το δούμε ε, σε διεθνές επίπεδο να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην Βουλγαρία οι μισοί χρήστες που χρησιμοποιούν του διαδικτύου βρίσκονται σε πάνω από 100 megabits per second και στόχος μας είναι να ανέβουμε ακόμη περισσότερο. Πρόκειται για εξελίξεις που είναι ε, σημαντικές. Στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι τεχνικά εφικτό, εφικτές μεγάλες ταχύτητες, αλλά αυτό είναι δαπανηρό. Αν μιλούμε λοιπόν στα σοβαρά για διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας, θα πρέπει να δαπανίσουμε και τα χρήματα. Μετά μιλάμε για οπτικές ίνες, και άλλα εργαλεία, άλλα μέσα διαβίβαση της πληροφορίας αν θέλετε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν παραδείγματα σε ορισμένε χώρες όπου το οπτικό δίκτυο είναι πάρα πολύ καλά ανεπτυγμένο. Αλλά σε γενικές γραμμές για την Ένωση δεν μπορούμε να πούμε ότι πετύχαμε και πολλά. Αν δεν χρησιμοποιήσουμε τα μέσα αυτά για την ε, μεταφορά δεδομένων ε, θα ειστερήσουμε και σε άλλες τεχνολογίες στο μέλλον. Έχουν γίνει πολλές και ενδιαφέρουσες συζητήσει και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα προϊόντα του διαδικτύου και κοινωνικής φύσεως στην Ευρώπη έχουμε ένα από αυτά τα προϊόντα, το Skype. Στις άλλες χώρες, στις Ηνωμένε Πολιτείε έχουμε το Facebook και άλλα τέτοια πολύ γνωστά προϊόντα, τα οποία δεν έχουμε στην Ευρώπη. Και έτσι η καινοτομία τρέχει περισσότερο στις άλλες χώρες και όχι στην Ευρώπη. Εγώ νομίζω ότι πρέπει πάρα πολύ σοβαρά και αυτό λέγεται βεβαίως και στην ε, έκθεση που θα ε, οριστικοποιηθεί σε λίγο εδώ στο Κοινοβούλιο. Αν θέλουμε να σκεφτούμε σοβαρά τα θέματα αυτά θα πρέπει να αρχίσουμε να θα παραδείγματο χάρη με ένα ε, είδος βιβλιοθήκης σαν το Google Library ε, που πρέπει να προωθήσουμε είδαμε τι έγινε τον τελευταίο καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την πρόσβαση στο Google θα πρέπει να είμαστε και γρήγοροι να βιαστούμε διότι εάν δεν βιαστούμε τότε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και οι εκδοτικοί οίκοι της Ευρώπης θα βρεθούν σε δύσκολη κατάσταση και όταν μιλάμε για κανονιστικές ρυθμίσεις στο διαδίκτυο σίγουρα δεν εννοούμε τον περιορισμό του διαδικτύου αυτό δεν μπορεί να γίνει υπάρχουν όμως θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, πνευματικά δικαιώματα ε, και τέτοιου είδους προβλήματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε για να δούμε πώς μπορούμε να τα λύσουμε λόγω της καινούρια κατάστασης στην, ε, των, των καινούριων συνθηκών στις οποίες ζούμε. Υπάρχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τώρα και η, ειδικά η κυρία Ρέντινγκ ε, ασχολείται και θα συνεχίσει να ασχολείται με την ε, ασφάλεια στο διαδίκτυο. Υπάρχουν τέτοιου είδους αρχές και τέτοιου είδους φορείς στην Ιαπωνία και αλλού στον κόσμο και νομίζω ότι σχετικά θα πρέπει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η δική μας Επιτροπή, να κάνει μια έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, όχι μόνο στο δίκτυο, στον κυβερνοχώρο. Αυτό που ονομάζουμε cyber security. Όταν μιλούμε λοιπόν για το μέλλον μας, ε, σε σχέση με το διαδίκτυο θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο φιλόδοξοι από ό,τι φαίνεται από αυτή την έκθεξη της Κομισιόν. Πρόεδρος, ευχαριστώ ιδιαίτερα. Είπατε πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές ιδέες. Ίσως μπορεί να σας απαντήσει ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα-πρώτα για τα σχόλια της συγκήτριας βεβαίως έχουμε συνέστηση της εργασίας που γίνεται και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και από τις Προεδρίες και από άλλους οργανισμούς είναι δύσκολο γίνεται πάρα πολλή δουλειά είναι δύσκολο να τις παρακολουθείς κανείς ε, όλες τις εργασίες αυτές αλλά τις ξέρουμε ότι γίνονται και ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη Σουηδική, Προεδρία, τη Σουηδική Προεδρία η οποία ε, έφτιαξε ένα κείμενο το Σεπτέμβρη με τίτλο Green Knowledge Society η πράσινη κοινωνία της γνώσης πάρα πολύ καλό κείμενο ε, έχουμε λοιπόν πληροφορίες και δεδομένα και πράγματι μπορούμε να σας δώσουμε και σας στοιχεία αν τα χρειάζεστε. Όσον αφορά τώρα τις προτεραιότητες και την ιεράρχησή τους, δεν μπορούμε ακόμη να πούμε ποιες θα είναι οι προτεραιότητες αυτές. Πρόκειται για πολιτική κρίση που πρέπει να γίνει ε, τώρα όσον αφορά τις δεξιότητες και τις ικανότητες σίγουρα είναι πολλές αυτές που απαιτούνται ε, πρακτικές δεξιότητες αλλά και ε, περαιτέρω ικανότητες και δεξιότητες αυτό που ονομάζουμε internet literacy για να μπορεί ο κόσμος να, ε, να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και να μαθαίνει αυτό μπορεί να το ξέρουν οι νέοι αλλά όχι οι πολίτες μεγαλύτερης ηλικία και ίσως δεν έχουμε ασχοληθεί α, αρκετά με το θέμα αυτό θα πρέπει να ασχοληθούμε γιατί σχετίζεται και με το θέμα της ανεργίας αυτό και τώρα μπαίνω στο θέμα της θέσης μας ε, παγκοσμίως αν δείτε την χρήση του διαδικτύου στην Ευρώπη και το συγκρίνεται αυτό με το τι γίνεται στην Αμερική. Βέβαια όλοι η νεολαία χρησιμοποιεί το ίντερνετ 80-90 ε, ε, τα 100 των νέων κάτω από τα, την ηλικία των 25 ετών χρησιμοποιούν το ίντερνετ, δεν το συζητούμε. στην Ευρώπη υπάρχει διαφορά ε, από τις από την ε, ε, Αμερική ε, και δεν ξέρω αυτό μπορεί να οφείλεται στη διαφορά μορφωτικού επίπεδου ε, η συμμετοχή ίσως ε, στα εργασιακά θέματα και τα λοιπά είναι επίσης διαφορετική στην Ευρώπη και στην Αμερική έχετε δίκιο λοιπόν πράγματι πρέπει να κάνουμε κάποιες συγκρίσεις και σε σχέση με το τι γίνεται διεθνώς. Ετέθηνα ερώτημα ε, γιατί στην Ευρώπη δεν υπάρχουν οι εταιρείε Web 2.0 που υπάρχουν στην Αμερική η απάντηση θα μπορούσε να σχετίζεται με τον κατακαιρματισμό και τη διαφορετικότητα των ε, κανόνων ε, και νομοθετικών ρυθμίσεων που διέπουν τις, την παροχή υπηρεσιών στο διαδίκτυο στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελείως διαφορετικές νομοθετικές διατάξεις στα 27 αυτά κράτη-μέλη ε, Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικές ρυθμίσεις, οπότε άμα ξεκινήσετε εσείς να παρέχετε υπηρεσίες στο διαδίκτυο μπορεί να ξέρετε τους κανόνες στην, ε, στη Βουλγαρία και μπορείτε ε, να μπορεί να είστε πολύ επιτυχείς στη χώρα σας, στη Βουλγαρία αλλά δεν ξέρετε τις, ε, την νομοθεσία στη διπλανή χώρα και το πιο εύκολο για σας θα ήταν να πάτε στην Αμερική να εκμεταλλευτείτε την ε, ε, αγορά των 300 εκατομμυρίων καταναλωτών αμέσως αντί να προσπαθείτε κομμάτι κομμάτι να ε, έρθετε σε επαφή με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης τα ασύρματα δίκτυα είναι και ε, το υλικό για τα σύρματα δίκτυα είναι πιο διαδεδομένο αλλού από ότι στην Ευρώπη αυτό είναι αλήθεια ε, τώρα οι βιβλιοθήκες και το Google στο οποίο αναφερθήκατε κοιτάξτε εδώ η Ευρώπη είναι πιο μπροστά από την Αμερική οφείλω να σας πω έχουμε πολύ καλύτερη ενημέρωση για τα πνευματικά δικαιώματα και συγγραφικά δικαιώματα κτλ. Μπορούμε λοιπόν να ξεπεράσουμε τις Ηνωμένε Πολιτείε αν υπάρξει συμφωνία για ορισμένα βασικά πράγματα και αν ε, ε, για, τα, για αυτούς που έχουν τις βιβλιοθήκες, για αυτούς που έχουν τα συγγραφικά δικαιώματα ε, και τα και κάποια τέτοια θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Από εκεί και πέρα ε, ξεκινήσαμε να κάνουμε μια τεράστια απογραφή, αν θέλετε, του, του, της κατά, του κεκτημένου αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Ποια είναι η κατάσταση. Πρόκειται για μια τεράστια μελέτη που φαζα, φαντάζεστε που αναθέσαμε σε μια νομική εταιρεία ε, και η οποία ελπίζουμε να μην αργήσει πολύ να τελειώσει ε, πρέπει να δούμε επίσης τι υπάρχει σε διεθνές επίπεδο γιατί ναι. υπάρχει μια διεθνή σύμβαση για το διαδίκτυο στην οποία όπως είναι μέλη μόνο 13 τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα τα οποία πρέπει ακόμη να τα δούμε Πρόεδρος ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι εδώ μπορούμε να κλείσουμε το θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης. Δεν βλέπω κανέναν άλλο να ζητεί το λόγο. Η συνάδελφος Δεκαστήλιο μας είπε ότι θα μας υποβάλει ε, τον Ιανουάριο μία έκθεση. Ε, Βέβαια είχαμε ορίσει μια ημερομηνία την 11η Ιανουαρίου, 11 Ιανουαρίου για καινούργια συζήτηση. Αυτό θα πρέπει να καταργηθεί γιατί έχουμε και την ακρόαση της Επιτρόπου ε, και θα δούμε μετά την υποβολή της έκθεσης πότε θα ξανασυζητήσουμε ε, το θέμα. Προχωρώ στο 14 επενδυτικά σχέδια σε ενεργειακή υποδομή. Δεν μπορούμε να αρχίσουμε ακόμη όμως γιατί η συγγήτρια κυρία Βάλεαν δεν έχει έρθει ακόμη. Έρχεται. Μη φύγετε ένα μικρό διάλειμμα ενός λεπτού.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 Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε με την ημερήσια διάταξη σημείο 14 επενδυτικά σχέδια σε ενεργειακή υποδομή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η συνάδελφος Βάλιαν είναι η συγκήτρια και έχει και το λόγο. Uh, Καλημέρα συνάδελφοι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη γιατί είδατε το σχέδιο έκθεσης και το επεξηγηματικό σημείωμα που παρουσιάσει καλά τα πράγματα. Είμαι ανοιχτή σε οποιασδήποτε ερωτήσεις και ιδέες και προτάσεις. Έχω όμως και κάποια σημεία, κάποια ζητήματα τα οποία θα ήθελα να συζητήσω περαιτέρω και με τους και και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλουμε να αυξήσουμε τη γραφειοκρατία και το διοικητικό φόρτο με αυτόν τον κανονισμό. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η Κομισιόν θα πρέπει να διευκρινίσει περαιτέρω ποιε είναι οι υποχρεώσεις ε, λογοδοσίας και υποβολής αναφορών και reporting ε, βάσει αυτής της διαδικασίας. Αυτό μπορεί να γίνει στον εφαρμοστικό κανονισμό της Κομισιόν. Δεν ξέρω όμω αν έχουν άλλε ιδέε και οι συνάδελφοι. Επίσης, νομίζω ότι θα πρέπει να διευκρινίσουμε περαιτέρω τα της ε, υποχρέωσης των επιχειρήσεων να κοινοποιούν επενδυτικά σχέδια ε, και πώς η υποχρέωση κοινοποίηση θα μειώσει το διοικητικό φόρτο όπως ισχυρίζεται η Κομισιόν θέλουμε να καταλάβουμε λιγάκι παραπάνω την φιλοσοφία τους, τη συλλογιστική της Κομισιόν σχετικά. Επίσης αναφέρεται το απόρριτο των ε, στοιχείων, ιδιαίτερα αν πρόκειται για εμπορικά στοιχεία, αυτό είναι πλήρως κατανοητό, αλλά υπάρχει, υπάρχουν κάποια θέματα που πρέπει να συζητήσουμε σχετικά. Η Κομισιόν προσπαθεί, ε, μάλλον πρέπει να διαχειρίζεται τα στοιχεία που παίρνει ουδέτερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό θα... και αμερόληπτα. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η κοινοποίηση αυτή καθεαυτή του επενδυτικού σχεδίου. Ε, εάν ζητείτε κοινοποίηση σε ένα αρχικό αρχικό στάδιο όπου δεν μπορούν να δοθούν πολλά στοιχεία. Τα πράγματα περιπλέκονται ε, και γι' αυτό θα ήθελα να ακούσω και άλλες απόψεις σχετικά. Όσον αφορά τώρα τον κατάλογο των σχεδίων, των projects που πρέπει να κοινοποιούνται ε, ε, αναφέρεται εδώ η εξόριξη πετρελαίου, φυσικού αερίου και τα λοιπά ε, και αναφέρονται κάποια κατόφλια ε, σχετικά με την υποχρέωση κοινοποίηση. Θα θέλαμε να τα συζητήσουμε αυτά. Και εδώ υπάρχει ένα σημαντικό θεσμικό θέμα. Τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας η οποία αναφέρει, έχει και το άρθρο 194 και όπου λέγεται ότι η ενεργειακή πολιτική υπόκειται στη διαδικασία της συναπόφασης λοιπόν ε, θα πρέπει να να δούμε ότι εδώ τώρα ζητεί η Κομισιόν να ενημερώνεται για όλα τα μελλοντικά επενδυτικά σχέδια για να έχει μια καθολική εικόνα της κατάστασης στην Ευρώπη. Αυτό είναι κομμάτι της ενεργειακής πολιτικής. Αλλά αυτά όλα είναι πράγματα τα οποία υπόκειται, επαναλαμβάνω, στη διαδικασία της συναπόφασης. Ε, ε, ε ζητώ εδώ γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών ε, Υποθέσεων ε, της Νομικής Επιτροπής του Κοινοβουλίου αυτό θα καθυστερήσει κάπως τα πράγματα αλλά είναι απαραίτητο να έχουμε τη νομική γνωμοδότηση ε, εν πάση περιπτώσει κλείνω εδώ και θα ήθελα να ακούσω την άποψη των συναδέλφων πρόεδρος ευχαριστώ πολύ ναι πρέπει να γραφεί και μια επιστολή σχετικά είχαμε συμφωνήσει για την επιστολή αυτή μετά άλλαξαν τα πράγματα τώρα θα τη γράψουμε την επιστολή αυτή βλέπω να ζητούν το λόγο διάφοροι συνάδελφοι Ο κύριος Μπάλσου διάβασα την, ε, το σχέδιο έκθεσης και είδα ότι υπάρχουν και πάρα πολλές τρόποι τροπολογίες. Υπάρχουν πολύ σημαντικές τροπολογίες μεταξύ αυτών. Ε, δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτές όμως, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο-τρία θέματα τα οποία για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ανάγκη βελτίωση του ανταγωνισμού και του ανταγωνιστικού κλίματος. Εκεί δεν έχουμε αντιρρήσεις. Ε, στον ενεργειακό τομέα βεβαίως υπάρχει ανταγωνισμός και βλέπουμε στην πρώτη τροπολογία να λέγεται ότι δεν πρέπει να υπάρχει επέμβαση στην αγορά. Ναι, ωραία, αλλά που μπαίνουν τα όρια αυτά τα οποία ζητείτε να μπουν εδώ. Άλλες αγορές για στερεοφωνικά παραδείγματο χάρη μπορεί να έχουν τους να ισχύουν κάποια πράγματα από αυτά που ζητούνται εδώ στις αγορές αυτές αλλά στην ενεργειακό τομέα χρειάζεται κρατική παρέμβαση και νομίζω ότι δεν μπορούμε να βάλουμε διαχωριστικές γραμμές και να πετούμε να μην υπάρχει ε, επέμβαση. Δεν θέλω τώρα να αποδηθώ σε έναν αγώνα κατά των αγορών, αλλά εδώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λιγάκι προσεκτικοί. Και είδαμε και με την ε, χρηματοπιστωτική κρίση ότι μπορεί κανείς να πρέπει να παρέμβει το κράτος, να παρέμβει σε ορισμένες περιπτώσεις. μην κάνουμε το ίδιο λάθος που είχαμε κάνει παλιότερα και εδώ. Πρώτο αυτό. Δεύτερο θέμα σχετικά με το απόρριτο των ε, δεδομένων που τονίζεται ιδιαίτερα στο σχέδιο έκθεση. Έχω την εντύπωση ότι εδώ υπερβάλλουμε λιγάκι και φοβάμαι ότι οι φορείς της αγοράς που και δίνουν δικά τους στοιχεία αλλά και χρειάζονται στοιχεία και ενημέρωση ε, δεν εξυπηρετούνται σωστά. Δεν πρέπει να παρα, εμποδιστεί η ροή πληροφοριών με το να τονίζουμε ιδιαίτερα την ανάγκη για το εμπόριτο των στοιχείων και την εμπιστευτικότητα. Ευχαριστώ πολύ ο συνάδελφος Κύρεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα έχω να σας πω την εξής παρατήρηση. Έχω προβληματιστεί πάρα πολύ όσον αφορά τους λόγους τις αιτίες, τα ελαττήρια για αυτόν τον κανονισμό γιατί ίσως θα ήταν πιο απλό το να προχωρήσουμε σε μια απόφαση του κανονισμού και έτσι να υπάρχει πλήρης πληροφόρηση. Όμως, νομίζω ότι τώρα προσπαθούμε να ενατενίσουμε το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. γιατί θέλουμε ασφάλεια ενεργειακή, θέλουμε ελληνική, θέλουμε επομένως συντονισμένη δράση από όλα τα κράτη-μέλη. Και έτσι να προχωρήσουμε σε κάποια έργα για την ενεργειακή πολιτική μα. Όμως αφού μιλάμε για αλληλεγγύη θα πρέπει να δούμε πώς θα ε, συμφιλιώσουμε, πώς θα γίνει συμβατή η ελληνική με την ανταγωνιστικότητα. Η Δε Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι χρειάζεται διαφάνεια. Όμως μας λέει ότι αυτά τα μέτρα δεν θα αφορούν την ε, πανευρωπαϊκή υποδομή για το μέλλον. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ε, ασάφεια. Και θα πρέπει να μην ξεχνούμε ότι επιβάλλεται να συνεργαστούμε. Θα πρέπει να έχουμε ένα κοινό όραμα, ένα κοινό πρόγραμμα για την υποδομή μας στο μέλλον. Ε, υγιής ανταγωνισμός αλλά και έλεγγυη. Δεν αποκλείει το ένα το άλλο. Επομένω, ο ισχυρός κανονισμός αλλά και ο κανονισμός τον οποίο τώρα συζητούμε θα πρέπει ακριβώς να εξυπηρετούν αυτό το σχήμα. Και φυσικά να εξυπηρετούν και οι πατριώτες των κρατών μελών. Άλλες παρατηρήσεις τώρα που έχω να σας υποβάλω είναι οι εξής. Αλλά έχω και κάποιες προτάσεις. Θα πρέπει πρώτα πρώτα να γίνει μια διάκριση. Έχουμε διαφορετικές διαδικασίες και διαφορετικές επενδύσεις σε σχέση με κάποιες άδειες που θα πρέπει να δοθούν τόσο ώστε να προχωρήσει μια επένδυση. Και πολλές φορές η άδεια της έγκρισης και της αδειοδότησης καθυστερεί τις ε, εξελίξεις. Έτσι δεν προχωράμε. Και επίσης είναι πάρα πολύ ενοχλητικό το ότι η διαδικασία από χώρα σε χώρα είναι διαφορετική. Πάντως, αφού μιλάμε για δίκτυα διαβίβασης, χρειάζονται ακόμη περισσότερες ε, άδειες η βιομηχανία πάντως δεν θα πρέπει απλώς να περιορίζεται σε χαμηλές εκπομπές, θα πρέπει να φροντίζει να είναι αποτελεσματική. Και αυτό γιατί η ασφάλεια η ενεργειακή αλλά και η παραγωγικότητα είναι οι προτεραιότητες. Για αυτή την πενταετία τώρα που έχουμε τάξει όσον αφορά την, τη μετατροπή, την ανανέωση των έργων υποδομής αυτό οπωσδήποτε μας οδηγεί σε αναγκαστικά σε, σε, προγραμματισμό. Να φροντίσουμε να έχουμε ενεργειακούς πόρους και για το μέλλον, εκτό από το παρόν. Οι δε εκπομπές του διοξιδίου δεν θα πρέπει να κατανέμονται ένα κλάδο, αλλά ανά εκπομπή μοναδιαία. Άρα έχει παραμέτρους ο κανονισμός αλλά δεν λέει πιο συγκεκριμένα τι παραμέτρους θα προβλέψει και δεν μιλώ για τις τεχνολογικές μόνο παραμέτρους. Δεν μιλούμε για πυρηνικά καύσιμα. Τα πυρηνικά καύσιμα θέλουν άλλου είδους συγκεκριμένα έργα υποδομής. Όπως τώρα την προσπάθεια που γίνεται για να υπάρξει κάποιο είδου αποθήκευση των πυρικών αποβλήτων. Αυτές οι παράμετροι που θέλουμε να τάξουμε δεν είναι τραπεζικά απόρριτα, θα πρέπει να είναι γνωστές σε όλους. Να εκπρόξουμε επομένω προς αυτό το περίφημο ανοιχτό σύστημα. Αλλά τι πάνε να πει ανοιχτό σύστημα και κλειστό σύστημα, δεν λέγεται αυτό. Όταν μιλούμε επίση για αποθήκευση. Αυτό ιδίω για τα ποινικά σημεία είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους ποινικούς σταθμούς του μέλλοντος. Θα πρέπει αυτό να είναι ξεκάθαρο. Επίσης η διασύνδεση δεν αναφέρεται παρά το ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο εάν θέλουμε να έχουμε τελικά μια αυθεντικά κοινή ευρωπαϊκή υποδομή. Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο του Ζαντού. Euh, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η πράσινη βεβαίως και συμφωνούμε με την εισηγήτρια για την νομική βάση. Και συμφωνούμε όσον αφορά αυτές τις γυμνές υποδομές που αναφέρει η εισηγήτρια. Το είπε και ο συνάδελφος Γκέρικ πριν από λίγο. Θα πρέπει όχι μόνο να πάμε προς ε, φυσικό αέριο και πετρέλαιο, αλλά να δούμε τι θα γίνει και με, την αποθήκευση ηλεκτρισμού και με όλα τα έργα υποδομής τα οποία καλύπτουν την ε, πυρηνική ενέργεια και όχι μόνο την παραγωγή. Συμφωνούμε με τις τροπολογίες της ηγήτριας για το κατόφλι και την ε, κοινοποίηση. Αυτές τα δέκα ΜΒ για την αιωλική ενέργεια είναι 40% της ε, παραγωγής αιωλικής ενέργειας. Τα ένα τέτοιο κατόφλι θα είχαμε μόνο 10% φωτοβολταϊκής ενέργειας που θα εκαλύπτεται και μόνο τη μισή παραγωγή γεωθερμικής ενέργειας. για να μπορέσουμε να καλύψουμε με αυτό το κατόφλι και άλλους ανανεώσιμους ενεργειακούς πόρους που ταχύως προχωράνε και αναπτύσσονται. Πάντως έχουμε κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά ε, το, το πόσο θα προβάλλονται αυτές τις προσπάθειες μέσω πρόθεσμα. Ε, λαμβάνουμε υπόψη αυτά που είπε η κυρία Βάλιαν, αλλά έχουμε μια μεριά την αξιοπιστία των στοιχείων, των δεδομένων και από την άλλη μεριά το, το το βασικό που είναι το να προλάβουμε τις μελλοντικές εξελίξεις. Άρα, όπως λέει η Κομισιόν, θα πρέπει να υπάρξει ένα, ένας καλύτερος τρόπος ε, λήψη αποφάσεων και όχι απλά ένα, ε, ένα, ένα μητρό που να περιλαμβάνει μόνο τα, τα κεκτημένα. Άρα χρειάζεται μία αντίστοιχη περίοδος κοινοποίησης και θεωρούμε ότι είναι σωστή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα για το διοξίδιο του άνθρακος, για τη συλλογή και αποθήκευση. Δεν λέμε τίποτα εδώ. Εξαιρείται η μεταφορά. Δεν ξέρω τώρα είναι θέμα διατύπωσης ή ουσίας. Η δε ε, εμπιστευτικότητα των δεδομένων όντως είναι κάτι το σημαντικό αλλά δεν ξέρω κατά, κατά πόσο αυτό λαμβάνει την υπόψη ότι πρόκειται για θέμα δημοκρατίας της ενέργειας για σήμερα και για το μέλλον. Άρα θα, το, το να, αναστεκόμαστε σε αυτό το απόρριτο τότε δεν είμαστε συνεπείς με το δημοκρατικό διάλογο που θα πρέπει να γίνεται. Άρα θα πρέπει να κάνουμε καλύτερη εξισορρόπηση μεταξύ αυτών των δύο, μεταξύ της διαφάνειας και του απόρριτου. κατακλείδη. Όντω θα πρέπει να γίνει γίνεται ευρύτερη διαβούλευση για την ανάλυση του τι θα ισχύσει για αυτό το κλάδο και ακόμα και αν δεν φτάνουμε στο κατόφλι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα τα εθνικά προγράμματα και ό,τι έχει σχέση με την αποκεντρωμένη ενέργεια να μπορέσει να καλυφθεί ούτω ώστε να μπορούμε να μην συνεπείς το στόχο μας για την παροχή και προσφορά ενέργειας. Να εξασφαλίσουμε επίσης ότι πολύ συχνά αναφέρεται στο κείμενο ότι δεν φτάνουμε στην επιθυμητή παραγωγή. Να διευκρινίζουμε αυτή την προσέγγιση ότι δεν πάμε από την ανεπαρκή στην υπερπαραγωγή. Και αν υπάρχει μια προσέγγιση που μπορεί πιο δυναμικά να καλύψει τη ζήτηση και τον στόχο της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας μέχρι το 2020, τότε θα μπορούμε να έχουμε σε μερικές περιπτώσεις τον κίνδυνο της ανεπαρκούς παραγωγής και αλλού τον κίνδυνο της υπερβολικής παραγωγής. Κάτι άλλο το οποίο δεν αναφέρεται στο σχέδιο κειμένου και είναι σημαντικό αφού θέλουμε να έχουμε μια ξεκάθαρη διαδικασία λήψη αποφάσεων για τις εγκαταστάσεις τότε θα πρέπει να, έχουμε, να ξέρουμε κάποια στοιχεία που αφορούν τη χρηματοδότηση γιατί σήμερα όλα τα ευρωπαϊκά κράτη αντιμετωπίζουν πρόβλημα όσον αφορά την κρατική χρηματοδότηση και για πολλά προγράμματα επιβάλλεται να είναι το δημόσιο που χρηματοδοτεί. Άρα θα πρέπει να προβλέπεται ε, και η ενημέρωση πληροφορία σχετικά με τη χρηματοδότηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ η Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την έκθεση. Νομίζω πως η κυρία Βαλεάν έκανε εξαιρετική εργασία και μας έδωσε μια εις εικόνα για την πρόταση. Μπορούμε να συμφωνήσουμε με τα περισσότερα στοιχεία από αυτά που προτείνει Έχουμε ωστόσο κάποια ανησυχία που αντικατοπτρίζεται σε κάποιες από τις δηλώσεις των συναδέλφων ε, εδώ, ιδιαίτερα νομίζω στις δηλώσεις του κ. Ζαντό και Γερή που αφορούν τις ε, τροπολογίες 9 και 10 της κυρίας Βαλεάν, οι οποίες προσπαθούν να συντομεύσουν το χρονικό διάστημα εντός του οποίου η επένδυση πρέπει να αναφερθεί. Και νομίζω πως εάν συντομευθεί αυτό, τη στιγμή δηλαδή που δίνεται η έγκριση για την επένδυση, τότε δεν γνωρίζουμε ακριβώς την κατάσταση. Ενώ ο στόχος μας είναι να, φωτίσουμε περισσότερο την ε, μελλοντική, το μελλοντικό σχεδιασμό των επενδύσεων. Δεν ξέρουμε, ας πούμε, ποια θα είναι η ακριβής κατάσταση για τον ηλεκτρισμό σε 10 χρόνια και γι' αυτό και προτείνουμε αυτό το όριο το πενταετές ε, πριν την επένδυση. Η φάση του σχεδιασμού προβλέπεται εδώ ακριβώς για να μας δώσει μια εικόνα για το πώς θα εξελιχθούν οι επενδύσεις στον ηλεκτρισμό αλλά και στους άλλους τομείς τα επόμενα 10-15 χρόνια. Αν δούμε μόνο στενά την ημερομηνία που ξεκινάει η δουλειά, ε, ε τότε ε, χάνουμε τις πιο μακροπρόθεσμες εξελίξεις. Γι' αυτό και είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά τις τροπολογίες 10 και 9 και είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη του κύριου Γκέρα και του κύριου Ζαντό που επίσης υπογράμμισαν τα συγκεκριμένα σημεία. Σε σχέση με την νομική βάση τώρα, έχουμε φυσικά διαβουλευτεί με την νομική μας υπηρεσία και μας είπε ότι υπάρχει λέξη specialis, ε, το άρθρο 373 και 187 της Ευρατόμ, της συνθήκης Ευρατόμ, 373 της συνθήκης Λισαβόνας και αυτά θα έπρεπε να εκλειφθούν ως νομική βάση και όχι το άρθρο 194 που αφορά την ενέργεια και αφορά την ουσία της πολιτικής. Φυσικά το συζητήσαμε αυτό και στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο μας ενημέρωσε ότι ήταν υπέρ του να ληφθεί υπόψη η οι τροπολογίες μάλλον του Κοινοβουλίου, αν και νομικώς δεν υποχρεώνονται να πράξουν κάτι τέτοιο. και θεωρούν ότι... Αλλά δεν είναι βέβαιοι ότι είναι το 337 η κατάλληλη νομική βάση. Ε, πάντως θα πρέπει νομίζω να συζητηθεί μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Για τα υπόλοιπα σημεία που αναφέρθηκαν υπάρχει κάτι το οποίο έχει προκύψει και στις δηλώσεις εδώ των συναδέλφων, δηλαδή η εμπιστευτικότητα των στοιχείων Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς στόχο έχουμε όχι να περιορίσουμε τη διαφάνεια, αλλά φυσικά βλέπουμε ότι τα εμπορικά κόστος ευαίσθητα στοιχεία θα πρέπει να προστατεύονται και αυτός και ήταν ο στόχος μας με αυτό εδώ το σχέδιο. Υπήρξαν κάποια αιτήματα να, από τον κύριο Ζαντό να συγκεντρωθούν άλλα στοιχεία, ιδιαίτερα αυτά που σχετίζονται με τα νοικοκυριά, αλλά νομίζω πως θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία σε σχέση με το φόρτο που θέλουμε να επιβάλλουμε στους ενδιαφερόμενους φορείς στα κράτη-μέλη από τη μια πλευρά και τη διαφάνεια που μπορούμε να πετύχουμε από την άλλη σε σχέση με τα νοικοκυριά. Ε, συγγνώμη, σε σχέση με τα νοικοκυριά νομίζω πως κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ εκτός αυτού του κανονισμού. Εμείς έχουμε έρθει σε επαφή με την Eurostat και μπορεί να συμπεριληφθεί η παραγωγή ηλεκτρισμού από τα νοικοκυριά στην επόμενη πενταετή τους έρευνα. Νομίζω πως αυτό θα ήταν ένας πιο σωστός τρόπος για να συλλέξουμε αυτά τα στοιχεία. Ο κύριος Γύρεκ είπε ότι δεν ε, ήταν πολύ ευχαριστημένος γιατί δεν εξετάζουμε πιο ουσιαστικά θέματα όπως το θέμα των εγκρίσεων, των αδειών και επίσης να δουλεύουμε με μια πανευρωπαϊκή υποδομή. Αυτό νομίζω ξεπερνά το πεδίο εφαρμογή αυτού του κανονισμού που περιορίζεται στη συλλογή πληροφοριών και όχι στην χάραξη πολιτικής. Όσον αφορά την Κομισιόν και την ε, πανευρωπαϊκή υποδομή, το χρόνο θα προετοιμάσουμε νέε κατευθυντήρε γραμμέ σε σχέση με τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργεια, όπου μπορεί να αναφερθεί και αυτό το θέμα, αλλά νομίζω πω ε, μάλλον θα ξεπερνά την πρόταση αυτή εδώ. Υπάρχει κάποια παρεξήγηση δε, έχω την εντύπωση, από τον κύριο Ντγκίρεκ και από τον κύριο Ζαντό σε σχέση με το ποια θέματα καλύπτονται Ίσως σε διμερείς επαφές θα μπορούσαμε αυτό να το διευκρινίσουμε. Λέει ο κύριος Γκύρακ ότι δεν καλύπτεται καθόλου η πυρηνική ενέργεια. Αυτό δεν είναι σωστό. Πρέπει να υπάρχει μια παρεξήγηση. Ιδιαίτερα γίνεται αναφορά στο παράρτημα στην πυρηνική παραγωγή, αλλά για την ε, ε, για τα πυρηνικά απόβλητα όντως δεν περιλαμβάνονται. Εκεί έχετε δει το ίδιο και για τον κύριο Ζαντό θα πρέπει να το κοιτάξουμε μαζί τα παραρτήματα. Επίσης θέλετε να καλυφθεί η χρηματοδότηση και πάλι αυτό ξεπερνά ε, το πεδίο εφαρμογή. Εμεί θέλουμε διαφάνεια όσον αφορά τι επενδύσει και πάλι υπάρχει και το θέμα της ουσίας σε σχέση με την απλή συλλογή στοιχείων. Γενικά είμαι ευχαριστημένος από τα σχόλιά σας. Ελπίζω πως θα ξανασκεφτείτε τι τροπολογίε 9 και 10, κυρία Βαλεάν, γιατί στην ουσία μα τραβάτε το χαλί κάτω από τα πόδια μας αν περιορίσετε το χρόνο παρατήρησης στην έναρξη της εργασίας και δεν συμπεριλάβετε το φάση του σχεδιασμού, γιατί ακριβώς αυτή είναι η ουσία της πρότασής μας. Πάντως σας ευχαριστούμε για τη γενική σας υποστήριξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Χιλμπρέχτ. Υπήρχε ένα θέμα νομικό. Ο κύριος Ροντρίγκες είναι εδώ από την νομική υπηρεσία. Ε, ίσως πρέπει να του δώσουμε το λόγο. Κύριε Ροντρίγκες, πρόεδρε. Πολύ σύντομα να σας δώσω μια πρώτη εκτίμηση όσον αφορά την νομική βάση. Όπως είπαμε, το 284 της συνθήκης ΕΟΚ ήταν το άρθρο επί, του οποίου ε, υποβλήθηκε η πρόταση αυτή στο Κοινοβούλιο. Τώρα, με την έναρξη ισχύω τη συνθήκη τη Λισαβόνα, υπάρχει, όπω ήδη υπόθηκε, το 194 η νομική βάση για την ενέργεια. Θεωρούμε ότι δεδομένου ότι βασικός στόχος αυτής της πρότασης είναι να συλλεγούν πληροφορίες ώστε να έχουμε και εδώ αναφέρω τη δεύτερη αιτιολογική σκέψη της πρότασης, ώστε να έχουμε μια γενική εικόνα της εξέλιξης των επενδύσεων στις υποδομές για την ενέργεια στην Ένωση. Δεδομένου λοιπόν ότι αυτό είναι ο κύριος στόχος αυτής της πρότασης, η νομική βάση του άρθρου 194 είναι η καταλληλότερη. Το γεγονός ότι αυτή η πρόταση αφορά την κοινοποίηση και τη συλλογή των στοιχείων, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι ο βασικό στόχο τη πρόταση. Ο βασικό στόχο είναι να συλλεγούν αυτά τα στοιχεία ώστε να έχουμε μια καλή εικόνα για την ενεργειακή αγορά και να διασφαλίσουμε τη σωστή τη λειτουργία. Στόχος που περιλαμβάνεται στο άρθρο 194 που είναι η νομική βάση για την ενέργεια. Γι' αυτό και θεωρούμε πως από αυτή τη νομική βάση θα πρέπει να ε, εξεταστεί αυτός, ε, αυτή η πρόταση. Τώρα για ένα άλλο θέμα, το γεγονός ότι υπάρχει η συνθήκη Ευρατόμ και η σχετική νομική βάση. Γιατί αυτή η πρόταση βασίζεται σε δύο νομικές βάσεις. Η μία είναι η συνθήκη ΟΚ, η άλλη είναι η συνθήκη Ευρατόμ. Για την Ευρατόμ βεβαίως γνωρίζουμε πως δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως η συναπόφαση και ε, αυτό σημαίνει πως η διάταξη αυτή της συνθήκης Ευρατόμ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση για αυτήν την πρόταση είναι το άρθρο 187 και μπορούμε να δούμε ότι μπορούμε να χωρίσουμε αυτόν τον κανονισμό. Από τη μια πλευρά έχουμε τον κοινοτικό νόμο άρθρο 194 με συναπόφαση και από την άλλη πλευρά, η κοινοποίηση επενδύσεων στις πυρηνικές εγκαταστάσεις ε, θα αντιμετωπιστεί με βάση το άρθρο 187 της Συνθήκης Ευρατόμ, δηλαδή απλή διαβούλευση του Κοινοβουλίου. Αυτή είναι η πρώτη μας αξιολόγηση και φυσικά είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω ε, πληροφορίες που μπορεί να χρειαστείτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο πρόεδρος. Θα πρότεινα και εγώ, όπως είπε και η κυρία Βάλιαν, να ε, φτιάξουμε μια επιστολή όπου να ζητούμε να μελετηθούν ορισμένα πράγματα και να ε, ζητήσουμε γνωμοδότηση νομική επ' αυτών όλων. Φαντάζομαι ότι ξέρετε τις, ε, <laughs> τις ημερομηνίες κατάθεση των τροπολογιών μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου και μετά το Γενάρη θα κάνουμε περαιτέρω συζητήσεις. Αν συμφωνείτε λοιπόν τώρα κυρίες και κύριοι, α, κύριε Χίλμπρεχτ θέλετε κάτι να πείτε Ναι ναι για την επιστολή ε, που είπατε ότι θα στείλετε Να τη στείλετε στην Κομισιόν Θα μπορείτε να στείλετε άλλη μια επιστολή την ίδια επιστολή και στο Συμβούλιο. Σωστό λέει ο Πρόεδρος. Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα να προτείνω κάτι επί της διαδικασίας γιατί έχουμε ένα πρόβλημα με την παρουσία κάποιων συναδέλφων. Αν συμφωνείτε θα θέλαμε να, προ... να συστήσουμε το σημείο 18 της κυρίας Ποδηματά. Απλώς μια παρα παρουσίαση της υπόθεσης θα μας κάνει η κυρία Ποδηματά να το συζητήσουμε τώρα και μετά να πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν κυρία Ποδηματά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ήθελα να σας ενημερώσω πολύ σύντομα για το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο και την Επιτροπή ε, γύρω από την οδηγία για τη σήμανση των προϊόντων που συνδέονται με την κατανάλωση ενέργειας στις 17 ε, Νοεμβρίου καταλήξαμε σε πολιτική συμφωνία με το συμβούλιο γύρω από το θέμα αυτό ήταν την ημέρα που ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις και γύρω από την οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων διεξήχθησαν συνολικά τρεις ε, ε, επίσημοι τρίλογοι και δύο τεχνικές συναντήσεις για τα επιμέρους ζητήματα που δεν είχαν ε, μείζωνα πολιτική σημασία. Ε, με δύο λόγια το τελικό αποτέλεσμα το αποτέλεσμα που αποτυπώνεται στην, ε, πολιτική συμφωνία ε, έχει ως εξής τα βασικά σημεία των διαπραγματεύσεων γύρω από τα οποία επικεντρώθηκε η συζήτηση η διαπραγμάτευση στους τριλόγους αφορούν στα εξής σημεία το πρώτο και σημαντικότερο όπως αντιλαμβάνεστε αφορά στη μορφή της ενεργειακής σήμανσης το περίφημο layout που ήταν και το πιο ε, αν θέλετε αμφιλεγόμενο το ζήτημα που προκάλεσε τις μεγαλύτερες αντιπαραθέσεις και τριβές ε, κατά τη διάρκεια της ε, σύνταξης του, αρχικού κειμένου μας και της διαδικασίας ψηφοφορίας σε πρώτη ανάγνωση. Αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο σημείο αφορούσε τις πρόνοιες για τις δημόσιες προμήθειες, τα κίνητα που θα πρέπει να χορηγούνται στους καταναλωτές αλλά και στη βιομηχανία για να ενθαρρύνονται να προάγονται τα περισσότερο ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα ε, οι διαφημίσεις των προϊόντων που συνδέονται με την κατανάλωση ενέργειας που καταναλώνουν ε, ενέργεια και το τελευταίο ε, αφορούσε τη διεύρυνση του στόχου της οδηγίας το αν και κατά πόσο δηλαδή θα φύγουμε από την στενή έννοια των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια και θα διευρύνουμε την ενεργειακή σήμανση και σε προϊόντα που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κατανάλωση ή αντίστοιχα στην εξοικονόμηση ενέργειας όπως επί παραδείγματι ε, τα υλικά οικοδομών τα κατασκευαστικά υλικά ε, που στο κείμενο που υιοθετήσαμε τον μάιο είχαμε ζητήσει να ενταχθούν ε, στους στόχους τους οποίους καλύπτει η συγκεκριμένη οδηγία. Ε, δύο λόγια λοιπόν για το τελικό αποτέλεσμα, για, τον, ε, ε, για την πολιτική συμφωνία στην οποία καταλήξαμε με το Συμβούλιο, αφού σας επισημάνω ότι κάτι που προφανώς γνωρίζετε ότι λόγω της θέσης σε ισχύ της συνθήκης της λισαβόνας αλλάζουν οι πρόνοιες που αφορούν στην επιτροπολογία στα delegated acts και στα implementing measures ε, και με αυτή την έννοια αυτά τα ζητήματα έχουν μείνει ε, ανοιχτά. Ε, ήδη περιμένουμε μια πρόταση από την επιτροπή στη διάρκεια αυτής ή και της επόμενης εβδομάδας. θα υπάρξει αντίστοιχη επεξεργασία από τη δική μας πλευρά από την πλευρά του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου στη βάση της οποίας θα διατυπώσουμε τις προτάσεις μας που θα πρέπει να ενσωματωθούν να ενταχθούν ε, στο κείμενο της οδηγίας για την ενεργειακή σήμανση. σε ό,τι αφορά στο αποτέλεσμα του διαλόγου πρώτα απ' όλα για τη σήμανση σας θυμίζω ότι σε πρώτη ανάγνωση είχαμε υποστηρίξει τη διατήρηση της κλειστής κλίμακας a 2 g με τακτικές αναθεωρήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα και την αναγραφή της ημερομηνίας διάρκειας της ενεργειακής ε, σήμανσης πάνω στο σήμα των προϊόντων. Ε, όπως ε, θα γνωρίζετε η μεγάλη πλειοψηφία των ε, αντιπροσωπιών στο Συμβούλιο αντιτάχθηκε σε αυτή την θέση και το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, των συζητήσεων που είχαμε με το Συμβούλιο αφορά στα εξής. Διατηρούμε την κλίμακα A to G με την δυνατότητα όταν η τεχνολογική πρόοδος το επιτάσσει να προσθέτουμε τρεις παραπάνω ε, τάξεις που θα αποτυπώνονται με τη μορφή του A+, A++, A++++, διατηρούμε τη χρωματική κλίμακα ε, έχει σήμερα με 7 ενεργειακές θέσεις και ταυτοχρόνως ε, υπάρχει πρόνοια επανεξέτασης της ε, ενεργειακής σήμανσης με σαφώς προσδιορισμένους όρους που περιγράφονται σε μια δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επισυνάπτεται ε, ε, στην, Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση. Σε ό,τι αφορά τις δημόσιες προμήθειες, σας θυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αρχική της πρόταση είχε ζητήσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε συμφωνήσει, είχε υποστηρίξει την υιοθέτηση διατάξεων για υποχρεωτικές ρυθμίσεις ό,τι αφορά στις δημόσιες προμήθειες. Ε, η θέση αυτή συνάντησε τη σφοδρή αντίδραση από την ε, πλευρά του, Συμβουλίου, παρά το γεγονός ότι ήταν ένα ζήτημα στο οποίο ε, δουλέψαμε μαζί και υποστηρίξαμε κοινέ θέσεις με την ευρωπαϊκή επιτροπή το τελικό αποτέλεσμα όπως αποτυπώνεται στο κείμενο της οδηγίας ε, αναφέρει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν ε, τις αρμόδιες αρχές την επισύναψη ε, συμβάσεων δημόσιων προμηθειών που θα προωθούν και θα επιλέγουν τα πιο ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα. τέλος σε ό,τι αφορά το, το θέμα της διεύρυνσης του στόχου της οδηγίας στα υλικά οικοδομών ε, συμφωνήθηκε να μην αποτυπώνεται ονομαστικά ο όρος υλικά οικοδομών μέσα στο κείμενο της οδηγίας αλλά να υπάρξει μια δήλωση ε, από την πλευρά της ευρωπαϊκής επιτροπής η οποία επίσης επισυνάπτεται στο κείμενο της οδηγίας με την οποία καθίσταται σαφές ε, ότι τα υλικά οικοδομών τα κατασκευαστικά υλικά καλύπτονται από το στόχο της οδηγίας για την ενεργειακή σήμανση και ότι η ευρωπαϊκή επιτροπή ε, αφού προχωρήσει σε μελέτες επιπτώσεων ανακατηγορία προϊόντων θα προτείνει εκεί ε, όπου πραγματικά κρίνεται σκόπιμο και ενδείκνυται ε, να συμπεριληφθούν τέτοιου είδους προϊόντα από, από τα εφαρμοστικά μέτρα της οδηγίας για την ενεργειακή σήμανση να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση τέλος ε, υπάρχει το θέμα των, διαφημίσεων των προϊόντων που συνδέονται με την κατανάλωση ενέργειας. Ε, στο, κείμενο που είχαμε υποστηρίξει σε πρώτη ανάγνωση τον περασμένο μάιο είχαμε ζητήσει ε, υποχρεωτική αναφορά στην ενεργειακή σήμανση ή στην κατανάλωση ενέργειας σε όλων των ειδών της διαφημίσεις προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια ήταν και αυτό ένα από τα σημεία αντιπαραθέσεων. Ε, μπορώ να πω ότι σε αυτό το θέμα ε, επικράτησε σε μεγάλο βαθμό η άποψη του Κοινοβουλίου καθότι στο τελικό κείμενο της συμφωνίας αναφέρεται με συγχωρείτε, ότι κάθε φορά που στις διαφημίσεις προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια υπάρχει αναφορά στην ενέργεια ε, ή στην τιμή του προϊόντος τότε υποχρεωτικά στη διαφήμιση αυτή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται αναφορά και στην ε, ενεργειακή σήμανση του προϊόντος. Αυτό ήταν σε γενικές γραμμές το, αποτέλεσμα. Ήταν μια δύσκολη ε, διαπραγμάτευση όπως δύσκολη ήταν και για την ε, οδηγία που αφορά στην ενεργειακή αποδοτικότητα των, των κτηρίων και με αυτά τα δεδομένα πρέπει να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα και με την ευκαιρία ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους σκιώδεις εισηγητές για τη βοήθειά τους τη γραμματεία ε, για την ε, πολύτιμη συμβολή της και την, ε, την ευρωπαϊκή επιτροπή. σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω ότι δύο ζήτησαν το λόγο. Σας παρακαλώ όμως να είστε πάρα πάρα πολύ σύντομοι. Ο κύριος Μπάλτσο. πέντε λεπτά eh, έχουμε κύριε Πρόεδρε. Ωραία λοιπόν τρεις ή λεπτά θα μπορούσα να μιλήσω τέλος πάντων. Λοιπόν, πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα ε, εδώ αν κατάλαβα καλά το, ε, υπήρξε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο μοιράστηκε στο κοινό και το κοινό δεν ξέρω κατά πόσον ενδιαφέρεται ή κατά πόσον πιστεύει ότι μπορούν να αποδώσουν μέτρα α, όπως η ενημέρωση για κάποια προϊόντα όμως πρέπει να αποδωσουν μετρα οπως η ενημερωση για καποια προιοντα ομως πρεπει να επιμεινουμε ε, η παρα παραγωγοί και κατασκευαστές θα πρέπει να επιμείνουν και σαν νέος ευρωβουλευτής προσπάθησα να ενημερωθώ και να ασχοληθώ λίγο παραπάνω με το θέμα. Ευχαριστώ την εισηγήτρια, ευχαριστώ και την Κομισιόν η οποία με βοήθησε να καταλάβω περί τίνος πρόκειται φοβούμε όμως ότι υπάρχουν ορισμένα πράγματα ε, για τα οποία δεν είχα ενημερωθεί παραδείγματος χάρη νομίζω ότι πέρασε από την Ολομέλεια μια, ένα θέμα για τα ψυγεία όπου η κλίμακα προς τα πάνω ήταν τελείως ανοιχτή δεν κατάλαβα καλά γιατί τώρα εδώ ακούμε ότι το νέο σύστημα θα έχει A+++ ε, κλπ κλπ ε, ίσως ε, ε αυτό το σύστημα θα είναι καλύτερο, θα υπάρχουν και νέες ετικέτες στα προϊόντα, αλλά εγώ νομίζω ότι κάτι τέτοιο με ένα όριο προς τα πάνω θα έπρεπε να ισχύει για όλα τα προϊόντα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο συνάδελφο Ρόντε. Εγώ θέλω απλά να πω, κυρία Αποδηματά, πω ε, βρίσκω πω κάνατε εξαίρετο έργο ε, γιατί είδα το ε, τελευταία πρόταση της Κομισιόν και ιδιαίτερα είδα και την πίεση από τα λιγότερο φιλόδοξα κράτη-μέλη και καταφέρατε μια, ένα συμβιβαστικό, μια συμβιβαστική λύση που είναι αξιοθαύμαστη. Συγχαρητήρια, κάνατε πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Σύντομα και επακριβή τα σχόλια και σημαντικές οι ευχαριστίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας και την κυρία Ποδηματά και να κλείσω το θέμα εδώ. Επανέρχομαι λοιπόν εντάχει ε, αμέσως στο σημείο 16 της ημερήσιας διάταξης είχαμε ζητήσει από την Επιτροπή να μας κάνει μια παρουσίαση σχετικά με τον κανονισμό για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος από τα επιβατικά αυτοκίνητα. Υπήρχαν πολλά ερωτηματικά, πολλές αμφιβολίες και γι' αυτό είχαμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει την παρουσίαση αυτή. Χαιρετίζω τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, τον κύριο και τον ζητώ να καθίσει πρώτα ο άνθρωπος και να του δώσω το λόγο να κάνει μια εισαγωγή. Ναι. Καλημέρα σε όλους. Λέγομαι Φίλιπ Αούεν, είμαι από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Θα ήθελα να ζητώ συγγνώμη που αναγκαστήκατε κάπως να αλλάξετε την ημερήσια διάταξη, τη σειρά των θεμάτων στην ημερήσια διάταξη σήμερα το πρωί για να με εξυπηρετήσετε. Θα ήθελα να μιλήσω ε, όπως είπε και ο πρόεδρος για τις εκπομπές ε, του διοξιδίου του άνθρακος υπάρχουν τρεις νομοθετικές πράξεις που σχετίζονται με τον κανονισμό για τις εκπομπές ε, και που θα παρθούν μέσω της επιτροπολογίας υπάρχει υπάρχει ας πούμε το άρθρο 11 για κάποιες εξαιρέσεις Υπάρχει το άρθρο 12 για την, τις ε, οικοκαινοτομίες, μεθοδολογία τη σχετική κτλ. Τους τελευταίους μήνες η Κομισιόν ε, όρισε για, αυτε, τις τρεις νομοθετικές πράξεις αυτές τρεις ομάδες εργασίας για να συζητήσουν ε, λύσεις για να μπορέσουν να εφαρμοστούν τα άρθρα αυτά. Επίσης έγινε και μια συνάντηση με τη βιομηχανία στις αρχές του Οκτωβρίου οχτώ συμμετέχοντες ε, μη κυβερνητικοί οργανισμοί κατασκευαστές ενός κατασκευαστών εκπρόσωποι των κρατών μελών κτλ. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θέσαμε το θέμα στη ε, στην κοινωνία και στη βιομηχανία και ακούσαμε τις απόψεις τους και τώρα προχωρούμε στον έλεγχο αν θέλετε για τις εκπομπές ε, του διοξιδίου του άνθρακος και για την προστασία αν θέλετε ή τις ειδικέ διαρρυθμίσεις για τους μικρούς κατασκευαστές ή κατασκευαστές ειδικών προϊόντων ελπίζουμε να προχωρήσουμε τα θέματα αυτά το Φεβρουάριο αλλά το τρίτο θέμα της οικοκαινοτομίας είναι σχετικά περίπλοκο και από άποψη αν θέλετε ε, ενιών και επειδή δεν είναι αρκετά όριμο το θέμα τώρα για τον έλεγχο των εκπομπών ε, το περιεχόμενο του σχετικού κειμένου αναφέρεται στις πηγές, στο ποιες αρχές είναι υπεύθυνε για να ε, καταγράψουν αν θέλετε τις εκπομπές από τα αυτοκίνητα, ε, πώς μπορούν να ε, πώ θα ενημερώνεται σχετικά η Κομισιόν, τι γίνεται με τα βιοκαύσιμα κτλ. Τώρα υπάρχουν και εξαιρέσει. Δεν η σχετική συζήτηση. Ε, αφορά στο ποιοι κατασκευαστές μπορούν να περιληφθούν στις εξαιρέσεις. Τώρα, η έννοια αυτή της οικοκαινοτομίας που ανέφερα προηγούμενα είναι πάρα πολύ ε, σημαντική. Προσπαθούμε να βρούμε έναν ορισμό, να ρωτήσουν, να δούμε ποιες είναι οι εφαρμογές, και θα μπορούσαν να είναι οι εφαρμογές. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση όσο έχει αυτή τη στιγμή. Δύο έγγραφα θα είναι έτοιμα στην αρχή της χρονιάς για την οικοκαινοτομία. Ε, αργότερα κατά τη διάρκεια του 2010 θα λάβετε ένα σχετικό έγγραφο. Πρόεδρος Ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν ξέρω για ποιες ομάδες εργασίας και επιτροπές μιλούσατε για την Επιτροπή Κλιματικών Αλλαγών. Δεν υπάρχει ακόμη αυτή η Επιτροπή. Ο κύριος Λάγκα ήμουν ε, εισηγητής για το θέματα αυτά της Επιτροπής Βιομηχανίας νομίζω ότι η επιβολή κανόνων είναι ο σημαντικό είναι ο τρόπος να λύσουμε το πρόβλημα παρόλο που υπάρχουν αντιρρήσεις το ίδιο και εδώ για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από τα αυτοκίνητα στην τελευταία έκθεση αυτοκινήτου στη Φραγκφούρτη είδαμε ότι παγκοσμίω όλοι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων προσπαθούν να επιτεθούν σε κάποιους κανόνες προσπαθήσαμε να επιβάλλουμε αλλά ε, παρόλα αυτά Άρα λοιπόν η επιβολή κανόνων ήταν ο σωστός τρόπος να προχωρήσουμε. Αυτή η επιβολή κανόνων ουσιαστικά ήταν αντίθετη προς αυτά που ήθελε η Κομισιόν τότε. Ε, η κυρία Αγγέλικα Νίμπλε ήταν, είχε λάβει μέρος στις διάφορες συζητήσεις που έγιναν ε, και η Κομισιόν ήταν αντίθετη όμως εμείς επιμείναμε και ε, μιλήσαμε και για την οικοοικονομία και καινοτομία με συγχωρείτε και είχαμε πει ότι μπλοκάρει τα πράγματα η Κομισιόν ανεφλογού. τέλος πάντων άλλαξαν τα πράγματα τώρα ε, υποβάλλονται καινούριε προτάσει προτάσεις της Κομισιόν ειδικά για τον έλεγχο των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος ε, τώρα είχαμε πει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ολόκληρο το όχημα ε. Ε, και εδώ παίζει ρόλο η οικοκαινοτομία αν πούμε ότι η καινοτομία ε, αναγνωρίζεται μόνο ε, αν και εφόσον ε, δίνεται χρόνος και έγκριση τύπου αυτά τα πράγματα όλα είναι τρικλοποδιές και τροχοπέδι στην πρόοδο το, ξανα, το είπα αυτό στην Κομισιόν παλιότερα το ξαναλέω ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος κυρία Νίμπλε συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο συνάδελφος Λάγκε. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω αυτά που είπε, υποστηρίζω αυτά που λέει, έχω τις ίδιες ακριβώς ανησυχίες. Ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής Βιομηχανίας τότε που ήταν εισηγητής ο κ. Λάγκερ και μέρο μέρος όλες αυτές τις τριμερείς ε, συζητήσεις που γίνονταν και ε, σε τελευταία ανάλυση ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αυτό το οποίο επέμεινε για τους, ε, τις ρυθμίσεις αυτές οι οποίες όμως πρέπει να εφαρμοστούν έτσι όπως τις φανταζόμαστε να πω και εγώ δύο λόγια για την οικοκοινοτομία σαν μέλος της Επιτροπής Βιομηχανίας βεβαίως ε, υποστηρίζω και εγώ την πρόθεση οικοκοινοτομιών και τις επενδύσεις ε, σε οικοκοινοτομίες αλλά όπως είπε και ο κύριος Λάγκερ η νησιών με πάει, ακολουθεί μια τελείως αντίστροφη πορεία από αυτή που θα θέλαμε εμείς δημιουργεί γραφειοκρατικά εμπόδια καθυστερεί ε, φρενάρει την πρόοδο και που δεν είναι λόγο λέω όπως είπε και ο κύριος Λάγκερ δεν ήταν αυτό το πνεύμα δεν μπορεί να είναι το πνεύμα αυτό της οικοκαινοτομίας και αυτόν που αποφάσισε το κοινοβουλίο ρωτώ ε, επίσης γιατί οι προμηθευτές εδώ δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως και οι κατασκευαστές δηλαδή γιατί πρέπει οι προμηθευτές να έχουν εγκρίσεις για κάθε ένα διαφορετικό τύπο και τα λοιπά και τα λοιπά και δεν μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τα πράγματα όπως κάνουμε για τους κατασκευαστές. Θα με ενδιαφέρε να ακούσω την άποψη της Κομισιόν. Οι προμηθευτές για επίσης γιατί δεν μπορούν να υποβάλουν ανεξάρτητα από κάποιο κατασκευαστή αίτηση για οικοκαινοτομία. Θα έπρεπε να μπορεί να γίνεται κάτι τέτοιο. Ο συνάδελφος Λάγκερ επίσης είπε ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί επιτρέπονται ε, οικονομίες τέλος πάντων ε, εγκρίνονται που επιφέρουν μείωση τουλάχιστον α, γιατί υπάρχει αυτό το κατόφλι του ενός γραμμαρίου ανά χιλιόμετρο δεν το καταλαβαίνω αυτό το κατόφλι είναι πάλι τροχοπέδι, εμπόδιο ή τρικλοποδιά θα έλεγα στην όλη υπόθεση. Παρακαλώ λοιπόν την Κομισιό να λάβετε υπόψη σας αυτά τα σχόλια και στο καινούριο έγγραφο που θα φτιάξετε. Εμείς θέλουμε να προωθήσουμε τις καινοτομίες και στην, στον τομέα του αυτοκινήτου και στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος αλλά δεν έχει κανείς το δικαίωμα να υπονομεύει ή να εμποδίζει την τεχνολογική πρόοδο ε, για πολιτικούς λόγους. Σας παρακαλώ να το λάβετε υπόψη σας και να το εφαρμόσετε αυτό. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος, ο συνάδελφος Έιλερ. Και εγώ θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια προς την ίδια κατεύθυνση. Ένα από τα βασικά εμπόδια που θέτει η Κομισιόν και η Γενική Διεύθυνση είναι ε, ε, αυτά που σχετίζονται με, και με την προθεσμία τη, το χρόνο των 12 μηνών ε, είναι τεράστιο χρονικό διάστημα αυτό για τις υπηρεσίες ελέγχου δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ε, ε, προσπαθούμε να μπλοκάρουμε τα πράγματα τεχνητά. Στη Γερμανία υπάρχουν και ιδιωτικοί οργανισμοί όπως το TÜV και άλλοι που μπορούν να κάνουν τον έλεγχο και μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν γιατί η Κομισιόν ε, τον ε, προβάλ, προτείνει τέτοιου είδου διατάξει και αν θέλει να προωθήσει την καινοτομία η Κομισιόν βάλει τουλάχιστον έξι μήνες αν θέλει να επιταχύνει τα πράγματα όχι δώδεκα μήνες δεν είναι βεβαίως ο, το βασικό, το μεγάλο χρονικό διάστημα του χρειάζεται η Κομισιόν για να ελέγξει ορισμένα πράγματα. Ε, αλλά είναι αδύνατον η Κομισιόν στα πλαίσια της επιτροπολογίας να χρειάζεται 12 μήνες συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ και θα ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Όουεν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει. Thank uh, Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις παρατηρήσεις. Νομίζω είπα εξ αρχής ότι βρισκόμαστε στο, στη φάση της ε, συζήτησης. Δεν έχουμε καν να συντάξει κάποιο νομοθετικό, και νομοθετική πρόταση αυτή τη στιγμή. Ακούμε τον κλάδο, ακούμε τα κρατημέλη, ε, είμαστε σε φάση διαβούλευσης, θα, θα συναντηθούμε με τους οργανώσεις των παραγωγών. Ε, υπάρχει ένα συνεχιζόμενος διάλογος σε αυτό το τομέα. Το θέμα για τους προμηθευτές που προέκυψε δύο φορές είναι σαφές. Ο κανονισμός είναι σαφής, η Κομισιόν το δέχεται. Πλώς θα πρέπει να ξέρουμε πόσο η καινοτομία θα εξοικονομήσει. Και αυτό είναι το θέμα. Γιατί οι καινοτομίες μπορεί να σχετίζονται με, τις, ε, με τον περιορισμό του διοξιδίου του άνθρακα μόνο όταν ξέρουμε σε ποια οχήματα έχουν τοποθετηθεί. Δεν μπορούμε διαφορετικά να το μετρήσουμε και σίγουρα συμπεριλαμβάνουμε τους παραγωγούς στο πεδίο εφαρμογή ε, του κανονισμού. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Τώρα το θέμα των 12 μηνών είναι σχετικά λογικό. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε περίπλοκα τεχνικά ζητήματα. Δεν έχουμε ιδέα ακριβώς ποια θα είναι όλα αυτά αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να κάνουμε κάποια αξιόπιστη αξιολόγηση όλων αυτών. Γιατί από τη μια η βιομηχανία μπορεί να θέλει αυτές τις καινοτομίες γρήγορα, όμως εμείς πρέπει να σκεφτούμε και, τους, και άλλες ε, ανθρώπους που θα προτιμούσαν η Κομισιόν όλα αυτά να τα ελέγξει πολύ προσεκτικά. Και δεδομένου ότι θέλουμε να έχουμε μια αξιόπιστη διαδικασία ελέγχου και επίσης επειδή υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία στην Κομισιόν που πρέπει να ακολουθηθεί μεταφράσεις και τα λοιπά, ε, νομίζω λοιπόν ότι 12 μήνες είναι ένα λογικό χρονικό διάστημα. Έπειτα, υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη που συμφωνούν προς ένα όριο και πάλι αυτό είναι ανοιχτό. Δεν έχουμε αποφασίσει, ούτε έχουμε κάνει πρόταση. Και πάλι σίγουρα υποστηρίζουμε την ιδέα του να προωθεί η τεχνολογία την καινοτομία, την καινοτομία στην ε, αυτοκινητοβιομηχανία και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε σε αυτό το τομέα. Επίσης το θέμα του ολόκληρου αυτοκινήτου θα πρέπει να υπάρχει ένας πλήρης κύκλος δοκιμών που να καλύπτει το ολοκληρωμένο αυτοκίνητο. Γιατί διαφορετικά μπορεί να γίνει μια έκθεση μέχρι να γίνει και η αναθεώρηση του κύκλου δοκιμών το 2014-2015. Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. Ο κύριος Λάγκερ, ναι, να κάνω μια πρόταση, να στείλουμε ένα ε, κείμενο με συγκεκριμένες ερωτήσεις προς την Κομισιόν για να μπορέσουν να συζητηθούν. Όχι, δεν χρειάζεται να στείλουμε κατάλογο των ερωτημάτων, λέει ο Πρόεδρος. Μπορούμε να στείλουμε μια επιστολή όμως προς την Κομισιόν που να λέει ποια είναι η γνώμη της Επιτροπής μας, της Επιτροπής μας επί της προτάσεως της Κομισιόν. Γιατί πραγματικά θέλουμε να βοηθήσουμε την Κομισιόν να επιτεχύνει τα πράγματα. Και νομίζω ότι έτσι θα πρέπει να προχωρήσουμε ε, υπάρχει σαφής απόφαση από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο είμαστε κομμάτι αν θέλετε της νομοθετικής αρχής ε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ε, ακούσαμε την άποψη της Επιτροπής θα φτιάξουμε την επιστολή θα τη στείλουμε στην Κομισιόν Λάγκαρ να ζητήσουμε όμως και από την Κομισιόν να μας δώσει απάντηση πριν από τις ακροάσεις των Επιτρόπων. Ωραία, θα το δοκιμάσουμε και αυτό λέει ο Πρόεδρος. Πολύ ωραία λοιπόν, είναι προφανές ότι θα το πω στην επιστολή μου. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ τον εκπρόσωπο της Κομισιόν για τις σύντομη, σύντομες απαντήσεις που έδωσε. βεβαίω συνεχίζονται οι συζητήσεις διότι όλοι είμαστε υπέρ της τεχνολογικής πρόοδου της καινοτομίας και της προσπάθειας να ξεπεράσουμε τις κλιματολογικές αλλαγές. Και τώρα κυρίε και κύριοι προχωρούμε στο αγαπημένο μου θέμα, το 19, τα διάφορα. Δεν έχουμε τίποτα για τα διάφορα. Πάω στο 20. Ε, αυτές οι δύο ημερομηνίε που αναφέρονται εδώ δεν ισχύουν διότι θα γίνουν οι ακροάσεις των επιτρόπων εκεί. Ε, στη δεύτερη ε, εβδομάδα του Ιανουαρίου θα συναντηθούμε βέβαια για τις ακροάσεις αυτές των ε, επιτρόπων το ίδιο και την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου χτες ελέγχθηκε τους συντονιστές ότι η γραμματεία θα φροντίσει να βρει καινούριε ημερομηνίε για να μπορέσουμε τέλο πάντων να συναντηθούμε κάποια στιγμή. Πάντω ευχαριστώ όλου του συναδέλφου σήμερα που δουλέψαμε τόσο καλά και μπορέσαμε να τελειώσουμε νωρί. Καλό είναι αυτό. Καλή σα μέρα.